Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής είπα της εκπροσώπου της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια σχετικά με την... τη Λιβύη ο υπουργό Τσέλεβιτς. Υπουργό Ντοφ Κυρία Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, σήμερα έχω την τιμή να εκπροσωπώ την κυρία Άστον η οποία σήμερα το απόγευμα ταξιδεύει προς την Μέση Ανατολή για να ετοιμάσει την ε, συνεδρίαση της επομένης εβδομάδας στον ΟΙΕ. Μου ανέθεσε λοιπόν να σας ενημερώσω σχετικά και να την ενημερώσω στη συνέχεια την ίδια. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποια είναι η δέσμευση της Πολωνίας για να βοηθήσει τη Λιβύη. Ήδη το Μάιο είχε πάει ο αρμόδιος υπουργός μας επίσκεψη στη Λιβύη. Πρόκειται, Πρέπει την Πρόκειται για μία φάση όπου ο Λιβικός λαός επέδειξε τεράστιο κουράγιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε τον αγώνα του Λιβικού λαού σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο σε πρώτη τη φάση δεύτερο στην φάση της ανθρωπιστικής βοήθειας κατά την κρίση και τρίτον είναι αυτή η τρίτη φάση με, για μετά την κρίση. Στάλθηκε ένα σαφέστατο μήνυμα στο καθεστώς ότι έπρεπε να γίνει σεβαστή η θέληση του λαού και ο δικτάτορας έπρεπε να φύγει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε προληπτικά μέτρα ούτε ώστε ούτε χρήματα ούτε όπλα να μπορούν να φτάσουν στον Καντάφη. Ο Καντάφη εγκατέλειψε την ε, Τρίπολη ε, και η βοήθεια επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών. Η ότι εκπρόσωπος συμμετείχανε σε πολλές συνεδριάσεις και στη Λιβύη και στο Κάιρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται για την ομάδα, με την ομάδα της Λιβύης που συνεδρίασε 1η Σεπτεμβρίου στο Παρίσι. Εμείς παρακολουθήσαμε με ιδιαίτερη αγωνία την πολιορκία της Μισράτα, την ε, ε, έλευση των προσφύγων στην ε, Τινησία και βοηθήσαμε όσο μπορεί, ρέσαμε με 52 εκατομμύρια ευρώ ε, ενίσχυση από την αρχή της κρίσης. Έχουμε ομάδες ε, στην Βενγάζη και στα σύνορα με την Τινησία και τώρα πια έχουμε και στην Τρίπολη. Μπορέσαμε να εκενώσουμε 24.000 4.000 άλλο δαπούς, κυρίως από τη Μισράτα και βοηθήσαμε τραυματίες, ε, συμβάλαμε στην προστασία του άμαχου πληθυσμού, στην ανθρωπιστική δράση κατά των ε, για, την ε, ε, εξάλληψη των ε, κάτε πήγουσα βοήθεια. Από τον Μάιο η κυρία Στον πήγε στην Βενγάζη και άνοιξε ένα γραφείο, εγγενίασε ένα γραφείο της Ένωσης που μας επέτρεψε να έχουμε άμεση επαφή με το Εθνικό Συμβούλιο Μεταπολίτευσης. Επίσης καταφέραμε να βρούμε περιοχές, ε, μη συγγνώμη, όπου μπορούμε να ενισχύσουμε άμεσα τον πληθυσμό ε, και, τον, ε, και τους πολιτικούς για την μεταπολίτευση. Το καθεστώς πλέον δεν υπάρχει. Ο Καντάφη και ο περίγυρός του πλέον έχουν φύγει. Εμείς παρακολουθούμε από κοντά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Εθνικού Συμβουλίου και των, και των πιστών του Καντάφη και προσπαθούμε να ε, παρέμβουμε για τη σταθεροποίηση της κατάστασης, να βοηθήσουμε για τον εκδημοκρατισμό, για τον αφοπλισμό, για την απόδοση δικαιοσύνης, για την ανάκαμψη της οικονομίας. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμα ε, μες οι επόμενες εβδομάδες. Να υποστηρίξουμε λοιπόν τη Λιβύη στο σεβασμό ορισμένων αρχών, στην ε, διασφάλιση του στενού συντονισμού μέσω του ΟΗΕ όλων των εταίρων διεθνώς. Θα πρέπει να μπορέσουν οι αρχές της Λιβύης να παρέχουν τις βασικές υπηρεσίες στον λιβικό λαό. Εργαζόμαστε και στις Βρυξέλλες και στη Νέα Υόρκη ούτως ώστε το χρήμα το οποίο έχουμε παγώσει στις τράπεζες να καταφέρουμε να το ξαναστείλουμε στη Λιβύη. Συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές του ΟΗΕ που ασχολούνται με την μεταπολεμική κατάσταση. Διαπιστώνουμε ποιοι είναι οι διάφοροι κρίσιμοι τομείς. Είναι σημαντικότατη η συνεργασία για να αποφύγουμε την επικάλυψη των διαφόρων προσπαθειών και να βοηθήσουμε τις λιβικές αρχές αυτήν τη φάση μεταπολίτευσης. Επίσης θα ήθελα να πω ότι κάναμε την πρώτη εκτίμηση μαζί με τους εταίρους μας στη Λιβύη. Αξιότιμη κυρίε, Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι τα πρώτα κείμενα τα οποία εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πραγματικά καθοριστικά για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών ιδεών και αυτό είναι καθοριστικό για μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στις πολιτικές ομάδες. Θα ξεκινήσουμε με το ΕΛΚ. Ο κύριος Σαλαφράγκα, έχετε τρία λεπτά. Κύριε Επίτροπε, εάν θεωρήσουμε ότι χρειάζονται έξι μήνες για να σταματήσει ένα δικτατορικό καθεστώς 40 ετών, αυτό το εξάμεινο είναι μια πολύ σύντομη περίοδος. Αν όμως κοιτάξουμε πόσες ζωές χάθηκαν και πόσο υποφέρει ο λαός της Λιβύης και πόσο θα υποφέρουν και οι επόμενες γενιές, η ανάλυση μας θα πρέπει να είναι λίγο πιο διαφορετική και βεβαίως πολλά πρέπει να γίνουν από τη στιγμή που καταραίει το καθεστώς Καντάφη. Η ανθρωπιστική βοήθεια, ο έλεγχος των συνόρων, η τάξη που πρέπει να επιβληθεί και αυτή η μεταβατική περίοδος η οποία θα είναι εξαιρετικά δύσκολη θα πρέπει να ακολουθείτε και από την έλλειψη ατιμορρησίας για όλα τα διαπραχθέντα εγκλήματα. Θεωρώ και εγώ ότι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χάρη στη δράση κάποιων κρατών μελών, και εδώ πρέπει να μιλήσουμε για τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, χάρη λοιπόν σε αυτή τη βοήθεια αλλά και στο θάρρος του λαού της Λιβύης μπορέσαμε να σταματήσουμε αυτό το αποτρόπιο καθεστώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε με αποτελεσματικότητα και με ταχύτητα θα έλεγα τους τελευταίους μήνες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ο πρώτο θεσμικό όργανο που αναγνώρισε το Συμβούλιο, το Μεταβατικό Συμβούλιο της ε, Λιβύης. Ήμασταν οι πρώτοι που το αναγνωρίσαμε. Στείλαμε 150 εκατομμύρια ανθρωπιστική βοήθεια και ανοίξαμε γραφεία στην Τρίπολη και Πιστεύω ότι το συντομότερο δυνατόν θα πρέπει να διορίσουμε και έναν επικεφαλής αντιπροσωπείας έτσι ώστε να μπορέσει να συντονίσει τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών επιτόπου. Επίσης, Ξέρουμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ζητήσει να ανοίξουν ένα γραφείο στην Λιβύη. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, γιορτάσαμε πριν από λίγες μέρες τα δέκα χρόνια από τις επιθέσεις ε, στη Νέα Υόρκη και πιστεύω πραγματικά ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να δείξουμε αξιοπρέπεια έναντι του αραβικού κόσμου, έναντι όλων αυτών που σήμερα κινητοποιούνται και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αφήσουμε ακραίες τάσεις Ισλαμιστές να επιδεινώσουν και να αμαυρίσουν την κατάσταση στις χώρες αυτές και να περιορίσουν με το φανατισμό τους την ελευθερία. Σας ευχαριστώ πολύ. Για τους σοσιαλιστές θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκόμες για τρία λεπτά. Είμαστε πολύ ευτυχείς γιατί βλέπουμε ότι μετά από 40 χρόνια δικτατορία και έξι μήνες πολέμου ο Καντάφη και το καθεστώ του μπορούν να δικαστούν. Πρέπει να δικαστούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από το Μάιο είναι παρούσα στη Λιβύη και πολύ σύντομα μπορεί να πει κανείς η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι παρούσα στη Λιβύη. Επίσης παγώσαμε και τα μέσα που, διαθέτουν, που διαθέτει το καθεστώς της Λιβύης παντού στον κόσμο. Έτσι ώστε αυτά να δοθούν στις ε, νέες αρχές της Λιβύης πρέπει να υπάρξει συντονισμός γιατί θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ακολουθήσουν μια εθνική πολιτική στη Λιβύη. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν συνοχής και συντονισμός και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σεβαστεί την αξιοπρέπεια και τη βούληση του λαού της Λιβύης. Πρέπει επίσης να επιτρέψουμε στα Ηνωμένα Έθνη να συντονίσουν την αστοπιστική βοήθεια και τη βοήθεια ανοικοδόμησης της Λιβύης. Πρέπει να στηρίξουμε τις προσπάθειες συμφιλίωσης, εδραίωσης του στρατού και ενσωμάτωσης των πολιτών που σήμερα είναι ένοπλοι στη Λιβύη στην κοινωνία των πολιτών. Θεωρούμε πραγματικά ότι η κοινωνία της Λιβύης χρειάζεται πολλές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά το συνταγματικό της δίκαιο αλλά και τον τομέα της ασφάλειας. Η αξιοπιστία της προσωρινής κυβέρνησης, της μεταβατικής κυβέρνησης, θα εξαρτηθεί από την υλοποίηση κάποιων βασικών αρχών, θεμελιωδών ελευθεριών και την εδραίωση ενός κράτους δικαίου. Πιστεύω ότι θα πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε και τους μετανάστες οι οποίοι υπέφεραν επί χρόνια και αδικαιολόγητα υπό το καθεστώς Καντάφη. Χαιρετίζουμε σήμερα τις δηλώσεις του κυρίου Τζαλίλη στην Τρίπολη που λέει ότι η Λιβύη θα είναι μια μουσουλμανική χώρα μετριοπαθής η οποία θα σέβεται το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ανθρώπινα των τα δικαιώματα των γυναικών και των μεταναστών. Και ελπίζουμε ότι η μεταβατική κυβέρνηση θα ξεκινήσει μια προσπάθεια συμφιλίωσης με τη συμμετοχή των νέων και των γυναικών σε όλους τους φορείς και οργανισμούς. Εμείς σαν Ευρωπαίοι θα πρέπει να λειτουργήσουμε σαν μια δύναμη που ήταν απούσα τόσα χρόνια. Η εξωτερική μας πολιτική έναντι του καθεστώτος Καντάφη ήταν μια πολιτική συμβάσεων, πετρέλαιο έναντι εξοπλισμού. Η νέα μας πολιτική θα πρέπει πραγματικά να σεβαστεί το λαό της Λιβύης και την ελευθερία και αξιοπρέπειά του. Ευχαριστούμε. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων, ο κύριος Όγιουλαν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ η κυρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφη έχει πάψει να υπάρχει στη Λιβύη, αλλά η χώρα βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση λόγω του εμφυλίου και αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα. Το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο ανέλαβε την ευθύνη να οικοδομήσει την ελεύθερη Λιβύη και πρέπει να γίνουν σεβαστές οι δημοκρατικές ιδέες από όλους. Η αποστολή αυτή είναι δύσκολη και νομίζω ότι και εμείς πρέπει να παίξουμε έναν πολύ σοβαρό ρόλο να υποστηρίξουμε την εφαρμογή της δημοκρατίας με όλα τα μέσα και να αντιταχθούμε σε οτιδήποτε την εμποδίζει. Μαζί με την ελεύθερη κοινωνία πρέπει να στηρίξουμε τη δημιουργία μιας φιλελεύθερης οικονομίας γιατί η οικονομική ανάκαμψη είναι βασική για να μπορέσει η χώρα να περάσει στη δημοκρατία. Γι' αυτό είμαστε υπέρ του ξεπαγώματος των λιβικών λογαριασμών και της άρσης των διαφόρων μέτρων αποκλεισμού και άλλων και κυρώσεων. Η στρατηγική οικονομική τομής πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του λιβικού λαού και η παραγωγή πετρελαίου και αερίου να συνεχιστεί, να ξαναρχίσει για να χρηματοδοτήσει τα καθήκοντα αυτά πρέπει να εγκαθιδρυθούν οι βάσεις ενός κράτους δικαίου γιατί και η ασφάλεια της χώρας απαιτεί δομές που να λειτουργούν. Από την εμπειρία της δικής μου χώρας της Εσθονίας δηλαδή μπορώ να σας πω ότι η οικοδόμηση των δημοκρατικών θεσμών μπορεί να χρειαστεί αρκετό χρόνο. Από τη μία χρειάζονται χρειάζεται υπομονή από την άλλη Πρέπει να έχουμε ένα όραμα για να βασίζεται η Λιβύη σε δημοκρατικές αρχές και σε βασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για τους πράσινους ο κύριος Κον Μπεντίτ για τέσσερα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Πρόεδροι, θα ήθελα να μιλήσω και για τη Λιβύη και για τη Συρία και για τη Μέση Ανατολή γενικότερα. Για τη Λιβύη τα πράγματα είναι πολύ απλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η τελευταία αντέδρασε σωστά αφού βέβαια δίστασε αρκετό καιρό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως υπόθηκε και προηγουμένως όθησε μάλιστα καλό αυτό την αναγνώριση του Μεταβατικού Συμβουλίου και σήμερα πρέπει να συνεχίσουμε την ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση και διάλογο με την νέα μεταβατική κυβέρνηση που θα οριστεί σε λίγο γιατί σήμερα και κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην Αίγυπτο και στη Λιβύη πρέπει να δούμε πώς θα οικοδομηθεί η Λιβύη του μέλλοντος. Είναι πολύ δύσκολο πρόβλημα. Όλοι θέλουν τη δημοκρατία αλλά είναι φανερό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει ένα θετικό ρόλο με οικονομική βοήθεια, επενδύσεις και τεχνική βοήθεια για να μην πω ιδεολογική η ανοικοδόμηση δηλαδή η οικοδόμηση μάλλον ενός κράτους που δεν υπάρχει βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολιτική έρημο υπάρχουν άτομα, πολεμιστές και μικρές απομονωμένες ομάδες εκεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο πολιτιστικό για την μετά τον πόλεμο περίοδο. Κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Πώς να αφοπλιστούν οι μαχητές, πώς να οικοδομηθεί η δημοκρατική κοινωνία. Και γι' αυτό πρέπει κάποτε το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν και το Συμβούλιο να κάνουν μία σε βάθος συζήτηση για την αποτυχία της πολιτικής μας τα πέντε τελευταία χρόνια γιατί οι σχέσεις μας οι συμφωνίες σύνδεσης με δικτατορίες είναι κάτι που πρέπει να το αναλύσουμε και να δούμε ποια είναι η ευθύνη μας προς τις χώρες αυτές. Για τη Συρία τώρα, το Κοινοβούλιο νομίζω ότι πρέπει να ξεπεράσει την απλή φάση των κυρώσεων, διότι στη Συρία το θέμα είναι ότι δεν πρόκειται μόνο για πετρέλαιο αλλά γενικότερα για υποθέσεις χρηματικές. Πρόκειται δηλαδή για μια περίπτωση που μοιάζει αρκετά με, τη νότια, με τις Νότιας Αφρικής. Πρέπει οι επιχειρηματίες να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να έχουν πια εμπιστοσύνη για το μέλλον τους στο οικονομικό, στον Άσαντ. Γι' αυτό Χρειάζονται μεν κυρώσεις για τις πεταλαϊκές εξαγωγές, όχι όμως μόνο αυτές. Δεν πρέπει να θέλουν να μπορούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να έχουν δοσοληψίες με τη Συρία. Τέλος για τη Μέση Ανατολή, η κυρία Άστον θα προσπαθήσει να πείσει τους Παλαιστινίους να μην ζητήσουν την αναγνώριση του κράτους των, στον ΟΙΕ Εδώ αναλαμβάνεται σοβαρές ευθύνες διότι σε όσους το λένε αυτό στους Παλαιστινίους, όσοι το λένε αυτό στους Παλαιστινίους πρέπει να τους πούνε και ποια είναι η εναλλακτική λύση. Διότι αυτή τη στιγμή δεν γίνονται διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ δεν διαπραγματεύεται. Αν θέλετε λοιπόν, και χρειάζεται εδώ προσοχή, τα δύο επόμενα χρόνια, ίσως τον έναν επόμενο χρόνο, θα δούμε μια ανάποδη διαδικασία να σημειώνεται στα κατεχόμενα. Δηλαδή η Παλαιστινιακή Αρχή θα δώσει το κλειδί στους Ισραηλινούς και θα τους πει ορίστε όλα αυτά Ισραήλ είναι, πέστε τα όπως θέλετε Ισραήλ και Παλαιστίνη αλλά να εφαρμόσουμε την απλή αρχή ο καθένας μία ψήφο. Το Ισραήλ φυσικά δεν θα δεχτεί γιατί η πλειοψηφία είναι Παλαιστίνη και θα θελήσει να δημιουργηθεί ένα κράτος με apartheid και μετά θα αναγκαστούμε να εφαρμόσουμε κυρώσεις κατά του Ισραήλ. Σήμερα λοιπόν το να παίρνουμε την ευθύνη να πούμε στους Παλαιστινίους περιμένετε δεν αρκεί. Πρέπει να τους πούμε περιμένουν γιατί. Εδώ και μήνες ολόκληρους ο κύριος Ομπάμα προσπαθεί και κανείς δεν κατόρθωσε να πείσει τους Ισραηλινούς να διαπραγματευτούν. Ο κύριος Λίμπερμαν, υπουργός εξωτερικών του Ισραήλ, δεν ξέρω τι μπορεί να δώσει στους Παλαιστινίους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τάνοκ για τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, οι δυνάμεις απελευθέρωσαν την Τρίπολη. Ξέρουμε όμως σήμερα ότι οι δυνάμεις ε, που πολέμησαν το καθεστώς Καντάφη έκαναν και διέπραξαν επίσης εγκλήματα, καθώς και αυτοί που πολεμούσαν ε, σαν μισθοφόροι για τον Καντάφη. Ξέρουμε σήμερα ότι αυτοί οι οποίοι καταπολέμησαν τον Καντάφη θέλουν να δημιουργήσουν μια δημοκρατία πολυκομματική, δεν ξέρω αν θα είναι δίκαιοι και ελεύθεροι αλλά όλοι ξέρουν ότι τα εγκλήματα που έγιναν δεν μπορούν να σβηστούν από τη μία μέρα στην άλλη. Η ομάδα μου βεβαίως στηρίζει το ΝΑΤΟ και θεωρούμε ότι μέχρι σήμερα ήταν πάρα πολύ καλή η δράση τους. Προστάτευσαν τους άμαχους, τους πολίτες της Λιβύης και ελπίζουμε ότι μετά από 40 χρόνια δικτατορία η διαδικασία εκδημοκρατισμού θα πρέπει να οδηγήσει σε πραγματικά ελεύθερες εκλογές και σε μια κυβέρνηση που θα εκλέξει ο λαός της Λιβύης. Θεωρώ ότι η αποχή της ε, Γερμανίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης είναι κάτι που έδειξε ότι χρειάζονται κάποιοι που παίρνουν πρωτοβουλίες, όπως ο πρόεδρος ε, Σαρκοζή, που πολύ νωρίς είπε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε το Συμβούλιο και θα πρέπει να βοηθήσουμε τη Λιβύη για την ανοικοδόμηση. Σήμερα ο πόλεμος ε, σκότωσε πολλούς από τους πολίτες της Λιβύης. Σήμερα πρέπει να βοηθήσουμε να ξαναδημιουργηθούν θεσμοί πολιτικοί και να ξαναδημιουργηθεί μια δημοκρατική κοινωνία στην Λιβύη. Να υπάρξει ασφάλεια και βασικές υπηρεσίες προς τους πολίτες της Λιβύης. Πολλοί κάτοικοι σήμερα της Τρίπολης δεν έχουν καν πόσιμο νερό, καθαρό νερό και θα πρέπει όλοι να αναγνωρίσουν τη μεταβατική κυβέρνηση στην Λιβύη καθότι ο πρώην φίλος του ο έχει φύγει από την εξουσία. Ξέρουμε επίσης ότι το πάγωμα των μέσων του καθεστώτος Καντάφη από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ακολουθηθεί από μια επιστροφή αυτών των χρημάτων και αυτών των αγαθών στη νέα κυβέρνηση για να μπορέσουν να ανοικοδομήσουν την Λιβύη. Ξέρουμε επίσης ότι τα δισεκατομμύρια που έκλεψε το καθεστώς Καντάφη κάποια στιγμή θα πρέπει να επιστραφούν στον λαό, χωρίς αυτό να οδηγήσει σε μία κατοχή από ξένα στρατεύματα. Οι γειτονικές χώρες όπως ο Νίγηρας οι οποίοι βοήθησαν ε, τον Καντάφη και οι οποίοι σήμερα υποψιαζόμαστε ότι κρύβουν κάποια άτομα του καθεστώτος, θα πρέπει επίσης να συνεργαστούν ε, με τη μεταβατική κυβέρνηση και βεβαίως να τιμωρηθούν όλοι, ακόμα και αυτοί που ήταν στην αντιπολίτευση, για τυχόν εγκλήματα πολέμου. Θέλουμε εδώ να χαιρετήσουμε όλους τους επαναστάτες, όλους τους εξαγερμένους, οι οποίοι βρήκαν το θάρρος να εξεγερθούν καθά αυτού του αποτρόπιου καθεστώτος. Θέλουμε επίσης να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες όλων αυτών που έχασαν τους δικούς τους που είχαν θύματα πολέμου. Ελπίζουμε όλοι να βρούμε μια δημοκρατική Λιβύη μετριοπαθή μουσουλμανική χωρίς καμία εξτρεμιστική και ακραία τάση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της ΓΚΟΥΕ ο κύριος Πόρτας για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Αραβική Άνοιξη είναι ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της χρονιάς. Γι' αυτό και προτείναμε να δοθεί το, το βραβείο Ζαχάροφ στην Αραβική Άνοιξη συμβολικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μας ήταν συνένοχες των δικτατορικών καθεστώτων ε, των χωρών στις ε, οποίες έγινε η Ευρωπαϊκή Άνοιξη, η Αραβική συγγνώμη Άνοιξη. Και λειτουργήσαν πάντοτε κατασταλτικά έναντι αυτών των χωρών με καταπολέμηση της μετανάστευσης, καταστολή κτλ. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Το ΝΑΤΟ με επικεφαλή στο Παρίσι και το Λονδίνο ξεπέρασαν κατά πολύ την εντολή που τους έδωσε ο ΙΕ και η δράση τους, ε, η βομβαρδιστική τους δράση συνεχίζεται παρά το, το ότι η κατάσταση έχει ηρεμήσει. Οι βόμβες του ΝΑΤΟ συνεχίζουν να πέφτουν και βομβαρδίζουν οτιδήποτε θα χρειαστεί αργότερα νοικοδόμηση. Η ανησυχία μου όμως πάει ακόμη πιο μακριά. Εγώ θα ήθελα το Εθνικό Συμβούλιο Μεταπολίτευσης να κρατήσει τις υποσχέσεις του για το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Κυρίως έναντι των γυναικών και των μεταναστών. Και η Ευρώπη πρέπει να υποστηρίξει αυτήν την αυτή τη θέση. Όλοι οι, οι ανοίξεις έχουν ως επακόλουθο τα φθινόπορα. Δείτε τι γίνεται σήμερα στην Τινησία και αλλού. Ε, και δεν είχαμε μόνο τον Καντάφη ή τα αεροπλάνα του ΝΑΤΟ που έσφαξαν κόσμο και οι επαναστατικές δυνάμεις προχώρησαν σε βιότητες. Η δημοκρατική αλλαγή πρέπει να είναι τίμια πρέπει ο λαός να αποφασίσει μόνος του. Δεν θα πρέπει να ανακατευτεί η Ευρώπη εφαρμόζοντας δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορούμε εμείς ε, να μποϊκοτάρουμε το, το πετρέλαιο από τη Συρία και να δεχόμαστε το πετρέλαιο από τη Γεμένη. Δεν μπορούμε να θελοτυφλούμε στο τι συμβαίνει στο Μπαχρέιν. Μόνο έτσι η Αραβική Άνοιξη θα μπορέσει να μην σταματήσει ποτέ. Εξ, ο κύριος Προβέρα, εξ ονόματος της ΕΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε μία ανακοίνωση της 5ης Οκτωβρίου η Επίτροπη Φιούλε και Μάλστρομ εξέφραζαν την ικανοποίησή τους για το διάλογο με την Τρίπολη και με μια ατζέντα που προέβλεπε την παναφρικανική πολιτική, διεθνή προστασία των προσφύγων, έλεγχο το, της μετανάστευσης. Αυτή η φιλόδοξη ημερήσια διάταξη διακόπηκε λόγω της αλλαγής καθεστώτος στην Τρίπολη. Το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τη Λιβύη για αυτά τα μεγάλα θέματα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την ενεργειακή προμήθεια. Αλλά ένα άλλο σημείο πολύ σημαντικό είναι η ενίσχυση της νέας λιβικής πολιτικής ηγεσία με ελεύθερες εκλογές που θα είναι και η πρώτη πράξη μιας μεγάλης διαδικασίας που θα οδηγήσει στην οικοδόμηση ενός σταθερού και δημοκρατικού κράτους. Το Η οικοδόμηση μιας δημοκρατίας είναι πολύ πιο δύσκολο πράγμα από ότι να κερδίζει κανείς ένα πόλεμο. Άμα δεν υπάρχουν δηλαδή μνήμες σε μια χώρα προηγουμένων δημοκρατιών. Θέλω ξέρω ποια συγκεκριμένα προγράμματα μπορούν να εφαρμοστούν σύντομα ώστε να μεσολαβήσουμε στην κοινωνία των πολιτών και πιο συγκεκριμένα στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης που αποτελούν τους πυλώνες για την πραγματική οικοδόμηση της δημοκρατίας τουλάχιστον στα κεφάλια των πολιτών. Μίλτσερ για 1,5 λεπτό από τους μη εγγεγραμμένους. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Βεβαίως και σε έναν τέτοιο πόλεμο υπάρχουν πολλές συνέπειες. Το θέμα είναι αν θα πετύχουμε να δημιουργήσουμε, να οικοδομήσουμε ένα δημοκρατικό σύστημα και πώς θα ξεπεραστεί το παρελθόν της χώρας αυτής. Οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει όπως παραδείγματος χάριν, δύσκολα γεγονότα του παρελθόντος πρέπει να ξεπεραστούν. Πάρτε το παράδειγμα στην Τουρκία με τη γενοκτονία των Αρμενίων. Πρέπει να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή να ξεπεράσει και να περάσει σε μία φάση συμφιλίωσης. Ξέρουμε επίσης ότι υπάρχουν πάρα πολλοί από τους πολίτες της χώρας αυτής που συνεχίζουν να είναι οπλισμένοι, πολύ νέοι, ενθουσιασμένοι, εξεγερμένοι που συνεχίζουν σήμερα να είναι οπλισμένοι. Τι θα γίνει αν αυτή η κοινωνία μπει σε τοπικές διαμάχες. Η περηφάνεια, η εθνική περηφάνεια των Λιβύων είναι κάτι που σήμερα υπάρχει. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί να μην εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση κάποιοι ακραίοι όπως Ισλαμιστές παραδείγματος χάρη. Και θα πρέπει να βοηθήσουμε τα χρήματα τα οποία διαθέτει η διεθνής κοινότητα σήμερα να χρησιμοποιηθούν με το σωστό τρόπο. Επίσης υπάρχει και το θέμα της ε, πετρελαϊκής παραγωγής, η οποία βεβαίως θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τους Λίβους με το καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ. Επόλοιποι ο κύριος Μπροκ για δύο λεπτά. Ε, πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι, κυρία Πρόεδρε, βεβαίω και είναι καλό νέο η πτώση ενό δικτατορικού καθεστώσεω. Μία καλή είδηση, ένα καλό μήνυμα που σήμερα μα οδηγεί στην ανάλυση ότι αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ΝΑΤΟ και σε κάποια από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι όλα. Από την άλλη μεριά, μια συντονισμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ακολουθήσει οι κυρώσεις μας οδήγησαν σήμερα στην ολοκλήρωση αυτής της επιτυχίας. Και σήμερα μπορούμε να εκτιμήσουμε τις συνέπειες αυτής της ε, επιτυχημένης πολιτικής. Η Λιβύη δεν μπορεί από μόνη της να ανταπεξέλθει. Πρέπει να τους στηρίξουμε και σε θέματα ανοικοδόμησης του δημοκρατικού καθεστώτος και σε θέματα κατάρτισης των νέων, την δημιουργία ενός νέου κόσμου στη Βόρεια Αφρική με εταιρικές σχέσεις και θα πρέπει να δούμε, και αυτό το λέω σαν προειδοποίηση στην Επιτροπή, τα χρήματα που δίνουμε να μην ανταποκρίνονται όπως το παρελθόν κατά 70-80% σε μελέτες, αλλά σε υλοποίηση προγραμμάτων. Αυτό περιμένουν οι άνθρωποι αυτής της περιοχές. Χρειάζονται ελευθερία και καλύτερες συνθήκες ζωής. Κυρίες και κύριοι, μια τελευταία παρατήρηση θα κάνω. Ξέρω θα μιλήσουμε για την Μέση Ανατολή λίγο αργότερα. Πρέπει να είμαστε υπέρ της δημιουργίας των δύο κρατών και τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει πραγματικά να ανοίξουν τη δυνατότητα για τους Παλαιστίνιους. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή θέσεων από μέρους του Ισραήλ, αλλά θεωρώ ότι η κυρία Άστον που σήμερα βρίσκεται στην Μέση Ανατολή θα πρέπει πραγματικά να βοηθήσει γιατί όλη η Ευρώπη αλλά ιδιαίτερα η χώρα μου έχουμε μία συγκεκριμένη αποστολή και ευθύνη προς την περιοχή αυτή και πρέπει να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για ένα καλύτερο μέλλον στην περιοχή. Ο κύριος Παντζέρη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Παραμένουν ακόμη ορισμένοι θύλακες αντίστασης του παλιού καθεστώτος και ακόμη και αν ε, ο Καντάφη γενικώ περιφέρεται και φοβάται το Εθνικό Συμβούλιο Μεταπολίτευσης ε, κάποια τελευταία κάποιους τελευταίους παραγμούς επιθέσεων. Νομίζω ότι πέρα από αυτά το πρόβλημα έχει λυθεί. Πρέπει να δούμε το θέμα ανθρωπιστικής βοήθειας, αφοπλισμού, παρεμβάσεις μέσω πρόθεσμες και μακροπρόθεσμες με ενίσχυση στην εκλογική διαδικασία κατά τη μεταβατική περίοδο, στην καπάση, στις θεσμικές capacity buildings και στην θεσμική εξέλιξη. Μετά από την κρίση που είδαμε είναι σωστό να λέμε ότι αυτή είναι η φάση ενίσχυσης του ρόλου της Ευρώπης με την, με την απαραίτητη αποφασιστικότητα. Εμείς δεν έχουμε μόνο ανθρωπιστική αποστολή και δεν έχω εδώ κατά νου μόνο τους μετανάστες που βρίσκονται στη Λιβύη. Εμείς δεν μπορούμε να λείπουμε από το τραπέζι που θα ορίζει το νέο γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής. Δείτε το νέο πρωταγωνιστή που έχουμε, την Τουρκία με την θριαμβευτική επίσκεψη του Ερντογκάν σε διάφορες αραβικές χώρες. Δεν μπορούμε εμείς να ε, ε, αναθέσουμε μόνο στις χώρες οι οποίες ε, συμμετείχαν στην αποστολή του ΝΑΤΟ την μεταπολεμική οργάνωση διότι όλα αυτά δεν μπορούν να οδηγήσουν σε πάντα σε καλά πράγματα. Διότι ξέρετε ότι για την οικοδόμηση της Νέας Λιβύης έχουμε και τα οικονομικά και ενεργειακά συμφέροντα. Και πέρα από αυτά δεν είναι ξεκάθαρο ποιο θα είναι το δημοκρατικό μέλλον της Λιβύης. Είναι πολύ σημαντικός λοιπόν ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η πορεία που έχουμε μπροστά μας δεν θα είναι ούτε απλή ούτε σύντομη και κυρίως εμείς θα πρέπει να έχουμε συνέστηση ότι δεν είναι προεξοφλημένος ο εκδημοκρατισμός. Ο κύριος Μακμίλαν Σκοτ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η απουσία της Λέδης Άστον είναι κάτι που με λυπεί. Απ' την άλλη αναγνωρίζω ότι έχει πιο σημαντικά πράγματα να κάνει την ίδια ώρα γενικότερα για τη διασφάλιση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, όπου όπως λέγεται συχνά έχει μειωθεί κατά πολύ από τις ε, δραματικές εξελίξεις στην Βόρεια Αφρική από την Αραβική. Θυμάμαι τι λέγαμε εδώ στην Ολομέλεια στις 8 νομίζω Μαρτίου όπου είχαμε ζητήσει πολύ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να αναγνωρίσει το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο Είχα την τιμή να είμαι από τους πρώτους Ευρωπαίους πολιτικούς που είχε καλωσορίσει τον Μαχμούτ Τζιμπρίλ, τον προσωρινό πρωθυπουργό, στο γραφείο μου τότε. Και η Βαρονέσα Άστον τότε δίσταζε να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη. Αυτό είναι κρίμα νομίζω γιατί μια πρωτοβουλία της Ευρώπης τότε θα είχε αποτέλεσμα. Αργότερα βέβαια αναγνωρίστηκε από τον Γάλλο πρόεδρο ο Τζιμπρίλ αλλά αυτό δείχνει τουλάχιστον ότι εδώ μέσα η αίθουσά μας έχει καταφέρει να κάνει ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Σε όλη την περιοχή οι εξελίξεις από την Αραβική Άνοιξη ε, εξελίσσονται άνισα. Έχω πάει στην Τινησία πρόσφατα όπου προβλέπονται σε λίγο εκλογές και θα ήθελα να πω στους συναδέλφους σήμερα και στους εκπροσώπους των άλλων θεσμικών οργάνων ότι πρέπει να είμαστε μεν έτοιμοι για αλλαγές αλλά και για αβεβαιότητα διότι το μέλλον δεν είναι τόσο καθαρό όσο ολομίζαμε πριν από μερικούς μήνες και καταλήγω λέγοντας ότι ελπίζω η Ολομέλεια να υποστηρίξει την πρόταση ε, το βραβείο Ζαχάροφ να δοθεί σε εκπροσώπους της Αραβικής Άνοιξης. Θα ήταν κάτι πολύ επίκαιρο και θα έδειχνε ότι ενδιαφερόμαστε για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και μάλιστα όχι μόνο στη Λιβύη, την Τινησία και την Αίγυπτο αλλά παντού στον αραβικό κόσμο. Ε, ευχαριστώ. Μπραντνερ για 1,5 λεπτό. Πιστεύω πραγματικά ότι τα επόμενα επίπεδα παρέμβασής μας θα είναι καθοριστικά. Οι επόμενες στιγμές, αν θέλετε, της ιστορίας της Λιβύης θα είναι καθοριστικές. Η ενοικοδόμηση, η δημιουργία καλύτερων συνθήκων ε, ζωής, η επιστροφή στις κανονικές συνθήκες, το πόσιμο νερό, και όλα αυτά θα πρέπει πραγματικά να τα κάνουμε μαζί. Και πέρα από την ανθρωπιστική βοήθεια υπάρχουν και κάποιοι άλλοι τομείς στους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε. Παραδείγματο χάρη να μεσολαβήσουμε στην συμφιλίωση, κάτι που είναι απαραίτητο μετά από μια τέτοια σύγκρουση και διαμάχη που έχει διαιρέσει την κοινωνία και το λαό της Λιβύης. Πρέπει επίσης από τη βία να περάσουν οι πολίτες της Λιβύης στην δικαιοσύνη, κράτος δικαίου, να προσφέρουμε ασφάλεια και μεταρρύθμιση. Και αυτό αποκοινού με όλους τους εταίρους περιφερειακούς και εταίρους της Λιβύης. Πρέπει επίσης να βοηθήσουμε όλους τους ε, οπλισμένους πολίτες της Λιβύης να επιστρέψουν στην κοινωνία των πολιτών και επειδή σήμερα υπάρχουν ευρωπαϊκές εταιρείες, συγκεκριμένα μία ευρωπαϊκή εταιρεία η οποία βρίσκεται στην Λιβύη και σκάβει και εκμεταλλεύεται τον ενεργειακό πλούτο της χώρας αυτής, θα πρέπει με μεγάλη διαφάνεια να δούμε πώς θα συνεχίσει αυτή η συνεργασία μεταξύ Λιβύης και δυτικών εταιριών. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο κύριος Κόβαλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε Επίτροπε, βλέποντας πώς εξελίσσεται η κατάσταση στη Λιβύη, νομίζω ότι ως Ένωση πρέπει να μιλήσουμε με ένα στόμα μια φωνή. Δυστυχώς δεν φαντάζομαι ότι δεν θα γίνει αυτό όμως. Τα πράγματα είναι σαφή, χρειάζεται να δοθεί ένα σαφές μήνυμα και προς τη Λιβύη και προς άλλες χώρες που έχουν πρόσφατα απελευθερωθεί από τις γνωστές εξεγέρσεις τους. Πρέπει να ενδιαφερθούμε ιδιαίτερα για την κοινωνία, για τους πολίτες των χωρών αυτών. Να προετοιμαστούν ελεύθερες εκλογές, δημοκρατία, όλα αυτά πετούν πολλή δουλειά και πολύ υποστήριξη από την Ένωση. Πρέπει να δώσουμε, είπα σαφές, μήνυμα ότι θέλουμε και είμαστε διατεθειμένοι να τους βοηθήσουμε, να τους δείξουμε το δρόμο που έχουν πάρει τόσο πολλές άλλες χώρες. Το η Βόρεια Αφρική πρέπει να τη δούμε σαν ένα σύνολο, να θυμηθούμε ξανά όλες τις διαδηλώσεις, τις εξεκέρσεις, τους νέους που ήθελαν ελευθερία, γιατί δεν έβλεπαν κανένα μέλλον στη χώρα τους και θεωρούσαν τον εαυτό τους, έβλεπαν τον εαυτό τους σαν κάτι ανεπιθύμητο από την κυβέρνηση. Πρέπει να γίνει καλή διαχείριση των υδάτων, να δοθούν νέες ευκαιρίες ώστε οι εξεγερμένοι αυτοί που διακινδύνευσαν τη ζωή τους να μην αισθανθούν τελικά ότι απογοητεύτηκαν και απέτυχαν και ότι δεν άλλαξε τίποτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευθύνη εδώ να στηρίξει τις ελπίδες τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Αγγουράκης. 1,5 λεπτό. Ο πόλεμος του ΝΑΤΟ κατά της Λιβύης κορυφώθηκε με τη σφαγή πολλών αμάχων στην Τρίπολη και άλλες πόλεις. Η πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση και ηπα με τους βομβαρδισμούς καθορίζει τις στρατιωτικές εξελίξεις και έτσι ευθύνεται απόλυτα για τα εγκλήματα αυτά. οι δυνάμεις των λεγόμενων αντικαθεστωτικών με ηγέτες πρώην συνεργάτες του καντάφη και με σημαία τη μοναρχία ολοκληρώνουν το καταστροφικό αυτό έργο. για μια άλλη φορά φάνηκε όμως η απίθμενη υποκρισία και βαρβαρότητα των κυβερνήσεων των ηπα και χωρών της ευρωπαϊκής Ένωση καθώς και ο ρόλος των διεθνών ιδιοσιογραφικών πρακτορείων που συμμετέχουν στην ιμπεριαλιστική προπαγάνδα ο στόχος του πολέμου δεν ήταν ο σύμμαχος των υπεριαλιστών καντάφη αλλά ο πλήρης έλεγχος από τις δυνάμεις του νάτο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε βάρος των αναγωνιστών τους. επιδιώκουν να εμπεδώσουν τη στρατηγική για τη νέα μέση ανατολή και να συντρίψουν τις λαϊκές εξεγέρσεις στη βόρεια αφρική και τη μέση ανατολή η απόφαση του συμβουλίου της ευρωπαϊκής ένωσης στις 1 η απριλη σχετικά με τη χερσαία στρατιωτική επιχείρηση της ευρωπαϊκής ένωσης στη λιβύη αποδεικνύει ότι οι κυβερνήσεις αναπτύσσουν όλο και περισσότερο ιμπεριαλιστική επιθετικότητα για να εξασφαλίσουν μερίδια προς όφελος των πολυεθνικών της ευρωπαϊκής ένωσης στη χώρα αυτή. οι δυνάμεις της υδροϋποταγής είναι εκτεθειμένες αφού στήριξαν τη δημιουργία ζώνης απαγόρευσης πτήσεων που αποτέλεσε τον προπομπό του δολοφονικού πολέμου χαιρετίζουν τώρα τη νίκη των αντικαθεστωτικών δηλαδή του νάτο και μιλούν για αλλαγή σελίδα στη λιβύη. τα παζάρια για τα πετρέλαια και την ανοικοδόμηση στη διάσκεψη των παρισίων δείχνουν ότι η μοναδική διέξοδο για του λαού είναι η πάλι ενάντια στον υπεριαλισμό, ενάντια στην ευρωπαϊκή ένωση και το νάτο ο δρόμο για μια άλλη κοινωνία για μια άλλη ανάπτυξη σε αυτή την περιοχή που μόνο αυτή μπορεί να εξασφαλίσει την ειρήνη και τη συνεργασία των λαών. Ευχαριστώ. Μπάτεν για μισή για ένα λεπτό. Δεν είναι στην αίθουσα ο κύριος Μάουρο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα κείμενο του ψηφίσματος που θα ψηφίσουμε αύριο για τη Λιβύη και πρόκειται για την παγράφραφο εκείνη που αφορά στην τοποθέτηση του κυρίου Τζαλίλ στην Τρίπολη και που λέει ότι η Λιβύη θέλει να είναι μια χώρα με μουσουλμανική, με τριοπαθής και το σύνταγμά της να το αντικατοπτρίζει αυτό. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για τη Λιβύη αλλά και για το μέλλον όλων των χωρών που δίνουν στην Μεσόγειο. Αυτό και για την Ινησία και για τις άλλες χώρες. Ρωτώ, τι κάνουμε εμείς, και το ρωτώ δηλαδή και στο Κοινοβούλιο, για να μπορέσουμε να είμαστε συνομιλητές όταν θα σε αυτήν τη διαδικασία όπου νέοι συνταγματικοί χαρτές θα ορίζουν τον τρόπο συμβίωσης εκατομμυρίων ατόμων. Το σύστημα είναι πάρα πολύ ε, ο Θεός βρίσκεται και στο Αμερικάνικο Σύνταγμα και σε εκείνο του Σουδάν. Αλλά η λειτουργία του Συντάγματος στους ΜΕΝ και στους ΔΕΝ διαφορετική. διαφορετική. Και οι Γάλλοι δεν έχουν στο Σύνταγμα τους το Θεό, ούτε οι Κινέζοι, αλλά και εκεί τα Συντάγματα λειτουργούν διαφορετικά μεταξύ τους. Προτείνω λοιπόν να έχουμε μία αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ας πούμε της Επιτροπής Θεσμικών Υποθέσεων ή της Επιτροπής που να μην πάει βέβαια να πει στους Λίβιους πώς να γράψουν το σύνταγμά τους αλλά να επαναλάβει στους Λίβιους αυτά τα οποία είναι οι πεποιηθήσεις μας και που αποτελούν θεμέλιο των συνταγμάτων μας και του τρόπου που εμείς ερμηνεύουμε τη δημοκρατία. Η κυρία De για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ έχω δει, είναι δύο πράγματα που συμμερίζομαι με τον κύριο Μάουρο και τον κύριο Πρόβερα. Το πρώτο για τη Σαριά και το δεύτερο για τη μετανάστευση. Μου είπανε ότι είχαμε την Ευρωπαϊκή Σημαία στην Τρίπολη, πολεμίζει, πολύ ωραία, αλλά η Επανάσταση ακόμη ανήκει στους Λίβιους. Και άμα εμεί θα πρέπει να ενισχύσουμε τη μεταβατική φάση, θα πρέπει να πάμε στο ψαχνό. Για το θέμα της Άρια που μας την ανακοινώνει ο Αμπτεζαλίλ θέλω να ξέρω κάτι παραπάνω τι θα πει η Σόφτα Σαριάτ τι θα... διότι το ένα καθεστώς ή το άλλο με το ίδιο σύνταγμα μπορεί να κάνουν ζημιές. Εμείς είδαμε Λίβιες, συναντήσαμε γυναίκες από τη Λιβύη, πάρα πολύ σημαντικές, ε, εκπληκτικές που μας είπαν ότι εμείς παλέψαμε χρόνια για να μπορούμε να συμμετέχουμε στις αποφασιστικές διαδικασίες. Τη μία μάλιστα την είχαν βιάσει κιόλας εκεί πέρα για όλες αυτές τις αγωνίστριες που θέλουν να συμμετέχουν στα τεκτενόμενα που θέλουν μια διαφορετική Λιβύη. Αυτό το συνταγματικό πλαίσιο δεν είναι λοιπόν περίεργο. Συμμερίζομαι λοιπόν εν μέρη την, την τοποθέτηση του κυρίου Μάουρο. Και ξαναθέτω το θέμα για τη μετανάστευση. Εγώ ήμουν η πρώτη που πολέμησε κατά τη συμφωνίας με τον Καντάφη για τη μετανάστευση σε μια χώρα η οποία παραβίαζε μεγαλοπρεπώς τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ξέραμε όλοι. Τώρα μου λέτε, εντάξει το πρόβλημα το έχουμε, έχουμε από εκεί όλη την υπόσαχάρια μετανάστευση που περνάει, είναι τεράστιο πρόβλημα. Αλλά μήπως ε, είναι δυνατόν να έχουμε μια άλλη άποψη, ένα άλλο όραμα για το πώς θα λύσουμε το πρόβλημα, να δούμε δηλαδή αυτή τη μετανάστευση πώς μπορούμε να την καναλιζάρουμε μέσα από ανάπτυξιακά προγράμματα, ας πούμε τώρα η Λιβύη χρειάζεται ε, μετανάστες για να ξαναχτίσει δηλαδή, Μήπως ε, μπορούμε να βρούμε άλλες ε, λύσεις πέρα από αυτά τα στρατόπεδα κράτησης στα οποία θα πηγαίνουμε για να δούμε αν περιφρουρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα ή όχι. Αυτά λοιπόν, αλλά με διαφορετική βλέπετε άποψη από τους άλλους, ερμηνεία μάλλον από τους άλλους. Λόχ Μπίλερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα η κατάσταση στη Λιβύη μας αφήνει την ελπίδη ότι στην εξουσία δεν θα είναι πια η αυθαιρεσία ενός προσώπου, αλλά θα υπάρξει ελευθερία στη Λιβύη με νέες δομές, κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζουμε επίσης να επικρατήσει το κράτος δικαίου, να δημιουργηθούν νέες τέτοιες αρχές και να υπάρξει ασφάλεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη νέα κατάσταση να εστιάσουμε την προσοχή μας στην οικοδόμηση αυτών των νέων θεσμών. Επίσης είναι επιθυμητό η, στη Λιβύη να επικρατήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να δημιουργηθεί ένα νέο καθεστώς και να επικρατήσει ένα νέο σύνταγμα. Είναι επίσης πολύ θετικό το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε να καταργηθεί η θανατική ποινή στην ε, Λιβύη και θα πρέπει να μπορέσουν και σε εμπόλεμη αλλά και σε ειρηνική κατάσταση να επικρατήσουν δημοκρατικές διαδικασίες. Είναι σημαντικό για την κοινωνία της Λιβύης να, υπάρξει, να υπάρξουν κυρώσεις και τιμωρία αυτών που διέπραξαν εγκλήματα πολέμου. Θα πρέπει να εμπνευστούμε από τα καλά παραδείγματα παρόμοιων καθεστώτων στην Λατινική Αμερική και το πώς οι κοινωνίες ανοικοδομήθηκαν και έγιναν δημοκρατικές μετά από χρόνια δικτατορίας. Ξέρουμε ότι η εμπόλεμη κατάσταση και εγκλήματα πολέμου μπορεί να δημιουργήσουν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και θα πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έγιναν και από τις δύο πλευρές κατά τη διάρκεια αυτών των συγκρούσεων και θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να αναλύσουμε την κατάσταση και να τιμωρηθούν οι υπέτοι. Ευχαριστώ κύριο Πρέντα για μισή λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τη Δευτέρα το απόγευμα Ζήτησα να μην είχαμε μόνο συζήτηση αλλά και ψήφισμα. Και το επιχείρημα μου ήταν ότι πολύ καλά να ψηφίζαμε πριν ξεφύγει ο Καντάφη ή τον πιάσουν εχμάλωτο. Διότι μέχρι την επόμενη Ολομέλεια Καντάφη δεν θα υπάρχει. Μετά από την πτώση του Γουαλίλα, η Λιβύη περνάει σε ένα καθεστώς μεταπολίτευσης που ελπίζουμε να είναι δημοκρατικό. Το είπαν και προλαλήσαντες ότι οι Λίβοι ξεκίνησαν όλη την ιστορία αλλά και τα ευρωπαϊκά κράτη έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε πολιτικό επίπεδο αλλά και επειδή ορισμένες από τις ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν μέσω του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό λοιπόν εμείς έχουμε ευθύνε σήμερα για την ανοικοδόμηση των δημοκρατικών θεσμών και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα με την παρατήρηση του κυρίου Μάριο Μάουρο. Αυτή η ενοικοδόμηση δεν θα μπορέσει όμως να ξεκινήσει όσο δεν επικρατεί η ασφάλεια. Χρειάζεται η εθνική συμφιλίωση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη Λιβύη. Πρέπει όμως να δικαστούν και οι ένοχοι, αλλά με δίκες δίκες. Ευχαριστώ κύριος Γκουαλτιέρη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μετά από 42 χρόνια δικτατορίας και 6 μήνες σειράξεων ήρθε η στιγμή της τροφής για τη Λιβύη προς τη δημοκρατία, την ειρήνη, την ανάπτυξη και αυτό το μέλλον βρίσκεται στα χέρια των Λιβύων και κανένας δεν μπορεί να διανοηθεί να τους επιβάλλει προ κατασκευασμένες λύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως έχει τεράστιες ευθύνες, αποτελεσματικό ρόλο να παίξει μέσα στην μεταπολίτευση. Μετά από την περιθωριοποίηση της ε, λόγω των ε, διαιρέσεων μεταξύ των μελών της ε, στην αρχή ε, της ε, επανάστασης και ενώ την υπόθεση την διαχειριζόταν σοφά θα έλεγα το ΝΑΤΟ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπόρεσε να δράσει και να, κατάφερε να συμβάλλει θετικά με το άνοιγμα του γραφείου στην Βενγάζη στην ε, Τρίπολη η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι εκεί η ΕΚΟ επίσης χρειάζεται τώρα μία ισχυρή πολιτική στρατηγική και αξιόπιστη να έχουμε ένα πολυμερές ισχυρό και αποτελεσματικό πλαίσιο ε, να μην έχουμε επικαλύψει στη δράση της διεθνούς κοινότητας ε, χωρίς ανταγωνισμούς και υποστήριξη στην μεταπολίτευση η οποία θα είναι μακρόχρονη και πολύπλοκη που θα πρέπει να στοχεύει στην εθνική συμφιλίωση χωρίς να υπάρχουν δηλαδή άλλες αιστείες διάσπασης στη χώρα και να διασφαλίζει την πρόοδο και τη δημοκρατία, να εγγυάται την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών, ανανέωση των ηθινών των τάξεων. Τα θέματα δημόσιας τάξης ε, ζητούν να αντιμετωπιστούν θέματα όπως είναι ο έλεγχος των συνόρων ή ε, το δικαστικό σύστημα, η ασφάλεια, έλεγχος του, του οπλισμού και της διακίνησής του, μια δημοκρατική roadmap, roadmap και μια συντακτική ε, πορεία. Πρόκειται για μια σημαντική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του και να υποστηρίξει όλη αυτή τη διαδικασία. Ε, ευχαριστώ. Ο κύριος Δανζόν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ ελπίζω ότι το ψήφισμα που θα ψηφίσουμε αύριο για τη Λιβύη και που είναι ιδιαίτερα συνενετική θα είναι εξίσου εύστοχη με αυτή που ψηφίσαμε πριν από έξι μήνες εδώ και όπου οι περισσότερες από, τις, ε, από όσα είχαμε προβλέψει, από τις διατάξεις που είχαμε προβλέψει ήταν σωστά. Καταδικάζαμε το καθεστώς Καντάφη, μιλούσαμε για την ευθύνη προστασίας ε, του αμάχου πληθυσμού, αναγνώριση της νομιμότητας του εθνικού ε, του μεταβατικού του Εθνικού Συμβουλίου και όλα αυτά αποτέλεσαν τη σπονδυλική στήλη της δράσης της διεθνούς κοινότητας. Πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμή σε όλες τις χώρες και κυρίως σε ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες δεσμεύτηκαν και διπλωματικά και στρατιωτικά για να βοηθήσουν τον λιβικό λαό στις εμπνεύσεις του για ελευθερία. Θα ήθελε επίσης να, να αποτείνω όρο τιμή στους πιλότους εκείνους που οι Γάλλοι είναι στις 19 ε, ε, του μηνός ε, βομβάρδιζαν τις εφοδιοπομπές του Καντάφη θυμίζοντας την παρέμβαση στη Βοσνία, Μπούκοβα ή Σρεμπρένιτσα. Οι προκλήσεις της μεταπολίτευσης είναι τεράστιες και δύσκολο και, και απέχουμε από την προσέγγιση των στόχων. Πρέπει να παίξουμε σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή τη φάση. Εμείς θα πρέπει να προτείνουμε βοήθεια και η υποστήριξη που να ξεπερνάει την ανθρωπιστική βοήθεια που δίνουμε σήμερα και να συνοδεύσουμε όλα τα κινήματα κοινωνίας πολιτών, ανασύσταση του συστήματος ασφάλειας και δικαιοσύνης και αυτό θα πρέπει να βασίζεται σε μία βασική αρχή ότι οι Λίβοι είναι αυτοί που θα πρέπει να ορίσουν τη μεταπολίτευσή τους και με τις καλύτερες προθέσεις του κόσμου δεν θα πρέπει εμείς να υποκατασταθούμε πούμε στις εμπνεύσεις του λιβικού λαού. Ευχαριστώ. Η κυρία Κοπά για ένα λεπτό. Στη Λιβύη η μάχη των δυνάμεων εναντίον του αυταρχικού καθεστώτος δείχνει να κερδίζεται οριστικά. Το καθεστώς Καντάφη μετά από μια μεγάλη αματοχυσία αποχώρησε. Σήμερα το μεγάλο ζητούμενο είναι η ανοικοδόμηση στη βάση της δημοκρατίας, της ισότητας αλλά και της ειρήνης η κατάσταση όμως είναι εξαιρετικά κρίσιμη ακόμα και χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται σε τραγικές συνθήκες χωρίς νερό φάρμακα και τρόφιμα. αν σε αυτό προσθεθούν τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες γίνεται σαφές ότι η ευρωπαϊκή ένωση έχει απόλυτο καθήκον να συνδράμει τη χώρα αυτή να σταθεί στα πόδια της. η ανθρωπιστική βοήθεια είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Όμω η οικοδόμηση ενό κράτου δικαίου δημοκρατικών θεσμών η αποφυγή δημιουργία ενό κενού εξουσία, αλλά και η συμφιλίωση είναι μεταξύ των μεγάλων προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ω ευρωπαϊκή ένωση. η ένωση δεν στάθηκε πάντως στο θέμα τη λιβύη στο ύψο των περιστάσεων. δεν τα κατάφερε να εκφραστεί με μια φωνή και επέτρεψε στο νατο να δείξει ότι είναι ο μόνο αξιόπιστο φορέα στον τομέα τη ασφάλεια σήμερα καλούμαστε να στηρίξουμε τη νέα λιβύη που γεννιέται και να εγγυηθούμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για ένα καλύτερο μέλλον του πληθυσμού της. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευτυχώ η αντιπολίτευση στη Λιβύη και με τη διεθνή βοήθεια κατάφερε να αντιμετωπίσει τη δικτατορία του Καβάφη. Τώρα πρέπει να τσιμπήσουμε τον συνταγματάρχη και να τον δικάσουμε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα κατά του λαού του. Το πιο σημαντικό όμως όλα αυτά είναι να επικεντρωθούμε στην ανοικοδόμηση της χώρας και να προσπαθήσουμε η Λιβύη να γίνει ένα κράτο, καταστεί κράτος δικαίου, δημοκρατική χώρα, να ξαναφτιάξουμε φτιάξουμε τις υποδομές, νερό, ηλεκτρικό, πετρέλαιο, δημόσια τάξη με αστυνομία και να μαζέψουμε όλα τα όπλα τα οποία κυκλοφορούν στην επικράτεια. Και όλα αυτά είναι τα ουσιαστικά στοιχεία για να πετύχουμε το για, για να βοηθήσουμε τη χώρα. Επίσης πρέπει να λύσουμε και το θέμα του Σαχέλ. Πρέπει τα σύνορα, ούτω ώστε να μην ξαναγυρίσουν πίσω οι μισθοφόροι. Θα πρέπει να επιτρέψουμε τη δημιουργία οργάνων που θα επιτρέψουν τον επαναπατρισμό των Λιβύων που έφυγαν ως πρόσφυγες. Πιστεύω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Ε, ευχαριστώ. κύριος Μπουσουτήλ για 1,5 λεπτό. Grazie President. Dak li seħ fil-Libja kienet ħolma li saret realtà u nixtieq nifraħ lil poplu. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον λαό της Λιβύης για την ανατροπή του καθεστώτος Καντάφη. Λυπάμαι βέβαια για την απώλεια πολλών ζωών, αλλά είμαι περήφανος και για το Κοινοβούλιο που ήταν από τα πρώτα διεθνή όργανα που υποστήριξε τη δημιουργία μιας ζώνης αεροπορικού αποκλεισμού. Τώρα βέβαια πρέπει να βοηθήσουμε τον λαό της Λιβύης να προοδεύσει, να κινηθεί προς το δρόμο της ειρήνης, της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Πρέπει να τον βοηθήσουμε να κινηθεί προς την ομαλότητα, να μπορέσει ο λαός αυτός να ζήσει κανονικά, να έχει την υγειονομική περίθαλψη που χρειάζεται, ηλεκτρισμό, νερό. Να βοηθήσουμε δηλαδή τη Λιβύη να οικοδομήσει δημοκρατικούς θεσμούς με κράτος δικαίου και τον διαχωρισμό των τριών εξουσιών. Έχουμε εμεί εμπειρία να τους διδάξουμε άμα χρειαστεί για το πώς δημιουργείται ένα δημοκρατικό περιβάλλον. Πρέπει να βοηθήσουμε, επαναλαμβάνω, τον λαό αυτόν. Ευχαριστώ, ο κύριος, η κυρία για ένα ο για λεπτό. Οι προθέσεις είναι καλές και έχουμε πολλές ελπίδες και ελπίζω ότι θα υλοποιηθούν όλα όσα έχουν γραφεί στο ψήφισμα και όλα θα γίνουν έργα πλέον στη Λιβύη. Πρέπει να πω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες αυτή τη φορά δεν δίφθηναν την ορχήστρα και η Ευρώπη ήταν ιδιαίτερα δυναμική η Ευρώπη τα κατάφερε και επίσης πρέπει να πούμε ότι η Ευρώπη δεν ήταν ενωμένη ευθύς εξ αρχής. Πρέπει όμως να καταδείξουμε την πραγματική μας ενότητα τώρα στη φάση οικοδόμησης ε, της δημοκρατίας ε, στη Λιβύη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι σταθερότητα δεν πετυχαίνουμε χωρίς δημοκρατία. Γι' αυτό λοιπόν είναι ουσιαστικό στο Λιβικό Σύνταγμα να υπογραμμίσουμε την σημασία της δημοκρατίας που θα αποτελεί θεμέλια λίθο της ε, νέας χώρας, της Λιβύης. Ο Καντάφη πρέπει να φύγει από τη χώρα ή να δικαστεί. η σχέση μεταξύ Λιβύης και Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην είναι μία σχέση ανταλλαγών, δηλαδή αποστολής πετρελαίου προς την Ευρώπη. Πρέπει να είναι μία ειλικρινή αμοιβαία σχέση. Και όπως έλεγε και ένας Πολωνός συνάδελφος που μόλις τώρα σκότωσα το όνομά του λέει ο μιλητής, πρέπει να έχουμε μία ελευθερία χωρίς τρόμο. Catch the Eye. Αντρική είναι, για ένα λεπτό. Και però Δεν είναι στην αίθουσα. Ο, Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλό είναι που έχουμε και ορισμένες καλές ειδήσει αυτή τη φορά. Είναι πολύ ευχάριστο ότι ο δικτάτορ Καντάφη εγκατέλειψε τη χώρα. Ε, δίνουμε πλήρη υποστήριξη στην εξέγερση στη χώρα αυτή και πρέπει να συνεχίσουμε να την υποστηρίζουμε. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σαρκόζη για τον ηγετικό ρόλο που έπαιξε στην υπόθεση αυτή. Τώρα όμως υπάρχει το μέλλον. Η Λιβύη έχει οικονομικούς πόρους και μπορεί να διασφαλίσει το μέλλον της. Και φυσικά έχει πετρέλαιο που μπορεί να διασφαλίσει το λαό της ένα καλό βιωτικό επίπεδο. Η Λέδη Άστον έχει σημαντικό ρόλο να παίξει για να υπάρξει σταθερότητα στη χώρα και δημοκρατική διακυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε το λόγο τώρα στην κυρία Νεντέλτσεβα. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Οι Λίβοι χρειάζονται μια καινούργια Λιβύη και γι' αυτό πρέπει να τελειώσει η ιστορία του Καντάφη αυτό το ματοβαμένο καθεστώς ε, δεν θα, δώσει, δεν θα τελειώσει παρά μόνο αν γνωρίζουμε πού βρίσκεται ο δικτάτορ και είναι ανίκανος να ξαναρχίσει τα ίδια. Ο, ένας σκληρός εμφύλιος πόλεμος διέρεσε τη χώρα και για να τελειώσει ένας εμφύλιος πόλεμος πρέπει να υπάρξει συμφιλίωση. Αυτό πρέπει να κάνει η Εθνική Μεταβατική Επιτροπή. Και η μετάβαση πρέπει να γίνει με ακριβοδίκαιο τρόπο. Πρέπει να δοθεί χρηματική βοήθεια αλλά και μεταφορά της δημοκρατικής μας τεχνογνωσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Νευντεβάλοβα. Σας ευχαριστώ. Η Λιβύη προς το παρόν βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Πριν από δύο εβδομάδες τα χρήματα επιχειρήσεων από τη Λιβύη απελευθερώθηκαν και συνεχίζουν να λειτουργούν. Πρέπει πραγματικά να επωφεληθούμε από προηγούμενες εμπειρίες και να βοηθήσουμε την ανοικοδόμηση της χώρας αυτής. Παραδείγματος χάρη είδαμε τι έγινε στο Ιράκ. Πρέπει να παρακολουθήσουμε την κατάσταση της Λιβύης πολύ προσεκτικά και να εμποδίσουμε περαιτέρω αιματοχυσία. Συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να ακούσουμε το λαό και να δώσουμε την εξουσία στο λαό. Είναι όμως μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, όχι μόνο για το λαό της Λιβύης, αλλά και για όλη τη διεθνή κοινότητα. Ευχαριστώ. Πάσκου. Μετά την πτώση της Τρίπολης είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στη Λιβύη και πολύ δύσκολη διαδικασία ενοικοδόμησης των δημοκρατικών θεσμών. Θα πρέπει να δούμε τι έγινε στο Ιράκ, γιατί όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να αποφύγουν περαιτέρω θύματα. Η συνέχιση της κατάστασης στη Λιβύη θα εξαρτηθεί πολύ από την τύχη του Καντάφη, ο συνεχίζει να είναι άφαντος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη δυσαρέσκεια και την βία που επικρατεί σήμερα στην κοινωνία, τη δυσαρέσκεια του λαού της Λιβύης. Διότι σήμερα αυτοί που κέρδισαν αυτόν τον πόλεμο ζητούν να υπάρξει μια πολυμερής διαδικασία και οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ σήμερα βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παρέμβουν στο παιχνίδι της εξουσίας στη Λιβύη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι η ανοικοδόμηση της Λιβύης από ό,τι ακούστηκε από όλους τους ομιλητές έχει την έννοια της ενίσχυσης της μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή με μία φωνή η Ευρώπη ολόκληρη θα πρέπει να βοηθήσει τους αραβικούς λαούς γενικότερα για να οικοδομήσουν τα νέα τους κράτη. αναμφίβολα αν δεν το πράξουμε εμείς αυτό θα υπάρξουν άλλα κράτη τα οποία θα επιτελέσουν ή θέλουν να επιτελέσουν αυτό το έργο. λαμβάνοντας υπόψη την τυχοδιοκτική στάση που τηρεί η τουρκία την οδιοκτικη σταση που τουρει η τουρκια σημερα στην ανατολική ευρώπη λαμβάνοντας υπόψη την ηγετική παρουσία της τουρκίας την προσπάθεια για ηγετική παρουσία της τουρκίας στη λιβύη θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η ευρωπαϊκή ένωση εάν θέλει να κρατήσει την τουρκία σε πορεία ένταξη στην ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να βοηθήσει αυτούς τους αραβικούς λαούς και ιδιαίτερα τη λιβύη ούτως ώστε να μην απομένει σαν μοναδικό παράδειγμα για τη λιβύη η τουρκία. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ. Οι επιπτώσεις της Αραβικής Άνοιξης έχουν, ε, διαφέρονται πλέον σε όλες τις πτυχές της εξωτερικής μας πολιτικής. Οι προκλήσεις είναι τεράστιες και όλα σήμερα μπορούν να γίνουν ανάπτυξη στη Λιβύη. Κοινή ανάπτυξη, συνεργασία, η οικονομική, η θεσμική, η ανθρωπιστική. Πρέπει να περάσουμε τώρα στην εφαρμογή. Η Ευρώπη μπορεί να υποστηριχθεί σε δύο μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή της για να συνοδεύσει αυτή την ανάπτυξη. Την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γυτνίαση και το Κοινοβούλιο της Ευρωμεσογειακής Ένωσης. Πρέπει να ενισχύσουμε αυτές τις δύο πολιτικές. Κυρίως το θέμα διασυνοριακής συνεργασίας που μας επιτρέπει να χρηματοδοτήσουμε συγκεκριμένα σχέδια επενδύσεις, κοινωνική συνοχή, περιβάλλον, κινητικότητα γύρω από τη Μεσόγειο. Κυρίως ευνοεί τη δημιουργία δικτύων τοπικής αυτοδίκησης που μπορούν να συνεργάζονται και ρεαλιστικά και ανάλογα με τις ανάγκες να επιτρέπουν στους πολίτες είναι αποδέκτες των ευρωπαϊκών ενισχύσεων. Ευχαριστώ. Σαρτζεντίνη τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πέρσι την ίδια εποχή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθούσε να ξεκαθαρίσει τι ήταν αυτά τα 60 εκατομμύρια ευρώ που είχε δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Λιβύη για την δράση και την προστασία των μεταναστών. Επρόκειτο ουσιαστικά για τον έλεγχο των συνόρων και για μετανάστες οι οποίοι ζούσαν στην υποχάρια περιοχή σε χώρες οι οποίες είχαν δικτατορικά καθεστώτα. Όλα τα άτομα αυτά έπρεπε να μην φτάσουν στην Ευρώπη. Βλέπουμε όμως ότι και στην Ερυθρέα και στην Αιθιοπία και στην Αίγυπτο και στο Σουδάν υπάρχει αυτό το φαινόμενο της μετανάστευσης. Ερωτώ λοιπόν την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Μπορείτε να μας εγγυηθείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα φτάσουν στην Ευρώπη. Θα ήθελα επίσης να ξέρω τι έγινε με τα 60 εκατομμύρια που θα δινόταν στη Λιβύη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εμείς έχουμε ιδιαίτερες ανησυχίες μετά από πέντε μήνες βομβαρδισμούς και εκατοντάδες αμάχους ε, που, που δολοφονήθηκαν και μια χώρα η οποία είναι ρήπιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα η οποία ε, που προκάλεσαν αυτοί οι οποίοι ήδη έχουν ξεκινήσει τη λαιλασία της χώρας και ετοιμάζονται να την ξαναχτίσουν. Θέλουν δηλαδή να ξαναχτίσουν ερήμην του λιβικού λαού αυτή τη χώρα, τη χώρα που κατέστρεψαν. Ο λιβικός λαός είναι το θύμα μίας κατάφορης παραβίασης του διεθνούς δικαίου. με πρόσχημα και υποκρισία ε, για να προστατεύσουν τους αμάχους τους βομβάρδισαν. Εμείς πρέπει να σταματήσουμε τον ευρωπαϊκό και αμερικάνικο εμπεριαλισμό. Οι λαοί πρέπει να αντιδράσουν παίρνοντας την τύχη τους στα χέρια τους. Σπάσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, στην κατάσταση αυτή δεν χρειάζονται περαιτέρω βομβαρδισμοί και εξοπλισμοί. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει στο εξή για το μέλλον της Λιβύης. Μέχρι τώρα ήταν αρκετά πλούσια χώρα και παρόλα αυτά εξαρτάται από τη βοήθεια και την υποστήριξή μας. Θα χρειαστεί να χορηγηθούν ακόμη και τρόφιμα στους πολίτες και να επιδιορθωθούν οι καταστροφές του πολέμου, τα σπίτια, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, να επανικοδομηθεί η δημόσια διοίκηση μετά από τον εμφύλιο. Πρέπει να γίνει η ανοικοδόμηση λοιπόν και να δώσουμε χείρα βοηθείας και εκτός από την ηλική πλευρά να χορηγήσουμε και να τους βοηθήσουμε και για την οικοδόμηση δημοκρατικών θεσμών ώστε να υπάρξει χρηστή διοίκηση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι θα είναι μακροχρόνια και μακρόπνοη η βοήθειά μας προς τους Λίβιους. Ο κύριος Όμπερ Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όντως η Λιβύη πρέπει να γίνει ένα κράτος δικαίου και δεν ξέρω αν η Θαρία είναι αυτό το οποίο θα βοηθήσει. Ακούσαμε πολύ προσεκτικά τον Μουσταφά Αλτζαλίλ, ο οποίος ζήτησε ένα μουσουλμανικό και μετριοπαθές καθεστώς. Σήμερα η Λιβύη είναι ελεύθερη χώρα χάρη στην παρέμβαση του ΝΑΤΟ και των δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε σήμερα ότι υπάρχουν σχέσεις μεταξύ του προηγούμενου καθεστώτος του Καντάφη και του κυρίου Σρέντερ, Σαρκοζή, Μπλερ και άλλων δυτικών ηγετών, οι οποίες δεν μπορούν να σβηστούν από τη μία μέρα στην άλλη. Εμείς βεβαίως θα πρέπει να στηρίξουμε την Λιβύη, να γίνει μια πραγματικά δημοκρατική και ελεύθερη κοινωνία, μια κοινωνία η οποία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η οποία μπορεί να ενσωματωθεί στην δυτική κοινωνία. είναι ο κύριος Μπρόνς. Δεν χρειάζεται να δέχεται κανείς να είναι υπέρ του Καντάφη για να αμφισβητεί τα κίνητρα της δύση για την παρέμβαση. η υποχρέωση πώληση του πετρελαίου με αντίτιμο χρυσό αντί για δολάρια το σχέδιο αυτό του Καντάφη είναι ίσως ο λόγος για τον οποίο το αντιτάχθηκαν. Πιστεύετε ότι με την ε, παρέμβαση αυτή η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαϊκή εταιρεία του κόσμου θα μονοπολίσει πια τα λιβικά πετρέλαια. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα για το κατά πόσον αυτό είναι θετικό ή αρνητικό, αλλά νομίζω ότι μπορεί να εξηγεί γιατί έγινε η παρέμβαση. Τον Επίτροπο Φιλε, εκ Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα έχω μια διπλή ειδονή. Πρώτον συμμετέχω στη συζήτηση αυτή που στην οποία συμμετείχε ο εκπρόσωπος της ε, ανωτάτης της υπάτης εκπροσώπου για τα εξωτερικά και από την άλλη η Κομισιόν και δεύτερον νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό τη συζήτηση αυτή να τη συγκρίνουμε και με προηγούμενες για ανάλογο θέμα για την ευημερία των χωρών της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και είναι σημαντικές οι εξελίξεις και οι αλλαγές από τότε μέχρι τώρα. Εκτιμώ ιδιαίτερα ότι από τη συζήτηση αυτή βγαίνει ένα στεναρό μήνυμα. Η Ένωση θα είναι αποφασισμένη να στηρίξει την καινούργια Λιβύη που να παίξει πλήρως το ρόλο της στον διεθνή και, και μεσογειακό χώρο. Δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω για τη βοήθεια που πρέπει να χορηγήσουμε. Πριν την πτώση της Τρυπόλεως είχαμε αρχίσει ήδη τη συνεργασία με την Εθνική Μεταβατική Επιτροπή μέσω της χορήγηση τεχνικής βοήθειας τεχνογνωσίας για την οικοδόμηση δημόσιας διοίκησης, στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του δημοκρατισμού μέτρα ανοικοδόμηση σχολείων και σχολικών προγραμμάτων και βοήθεια προς μετανάστες και εκτοπισμένους. Τώρα, η κατάσταση στη Λιβύη έχει αλλάξει από τότε που έπεσε η Τρίπολη στα τέλη Αυγούστου. Την 1η Σεπτεμβρίου διεθνής διάσκεψη αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων καθώς και πρόσωποι διεθνών οργανισμών με, συναντήθηκαν με το, την Εθνική Μεταβατική Επιτροπή στο Παρίσι και όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τη στήριξή τους προς την καινούργια Λιβύη. Την επόμενη μέρα 2 Σεπτεμβρίου ζητήθηκε ο καθορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων για το έργο της Εθνικής Μεταβατικής Επιτροπής ώστε να χορηγηθούν τα υπεσχημένα. Ο πρόεδρος Μπαρόσο παρίστατο και μαζί με άλλους με το έγγραφο «Ανταπόκριση στην πρόκληση της σταθεροποίησης της Λιβύης» έδειξε καθώς και με άλλο έγγραφο της Κομισιόν που αφορούσε και αυτό τη σταθεροποίηση ότι υπόσχεται η Κομισιόν την στήριξη της διαδικασίας αυτής σταθεροποίησης της Λιβύης. Επίσης ακούστηκαν μηνύματα του, της Εθνικής Μεταβατικής Επιτροπής για τον τρόπο με τον οποίο οι δωρητές θα χορηγούσαν τη βοήθειά τους τόσο η Ένωση όσο και η Παγκόσμια Τράπεζα με πραγματιστική προσέγγιση του καθορισμού των πραγματικών αναγκών της Λιβύης. Σε αυτή τη δεύτερη μέρα της διάσκεψης η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε επίσης συμφωνίες για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, των γυναικών, τη διαχείριση των υδάτων την ελευθεροτυπία και άλλα. Αυτά με πλήρη υποστήριξη των νέων λιβικών αρχών προσωρινών. Μία, η κοινή υπηρεσία εξωτερικών δράσεων δηλαδή προετοίμασε αρκετά την ε, περιγραφή που πρέπει να κάνει, η λεπτομερή περιγραφή των αναγκών της Λιβύης τη αιτήση των αρχών της Λιβύης ζητήθηκε περισσότερη, ζητήθηκαν περισσότερες μελέτες και μεταφορά τεχνογνωσίας και εμείς ήδη επεξεργαζόμαστε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα χρηματοδότης της Λιβύης 11 με 13 σε ύψος 60 καταρχάς εκατομμυρίων σύμφωνα με τις ανάγκες που καθόρισαν οι Λιβικές αρχές. ανάγκες βέβαια που είναι υψηλότερες από αυτές που μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε αυτή τη στιγμή. Κατά, της, κατά τη σημερινή συζήτηση σημείωσα πολλές προτάσεις που ακούστηκαν παραδείγματος χάρη από την κυρία Μπραντνερ για τη συμφιλίωση ώστε ε, για την ε, τιμωρία όλων όσων έχουν διαπράξει βιοπραγίες για τον καθορισμό μιας νέας δεοντολογίας για την αναδόμηση της Λιβύης καθώς και τις προτάσεις της κυρίας Ντεκέιζερ για την ανάγκη να εξεταστεί και η μετανάστευση, η μετανάστευση από διαφορετική οπτική γωνία από ό,τι μέχρι τώρα. Αυτά τα θα τα εξετάσω σοβαρά, θα τα μεταφέρω στους συναδέλφους μου δεόντως. Τέλος, η Λιβύη έχει πόρους. Το ξεπάγωμα των λιβικών λογαριασμών θα επιτρέψει να αρχίσει ήδη η ανοικοδόμηση αλλά πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ένα σταθερό πλαίσιο για τη διαχείριση των πόρων, των πετρελαϊκών πόρων και του φυσικού αερίου. Και μετά η Κομισιόν θεωρεί ότι θα πρέπει να τεθεί κατάλληλη βάση για πιο μακροπρόθεσμες σχέσεις με την καινούργια Λιβύη. Είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε συμφωνία με τη Λιβύη του ίδιου τύπου με άλλες ε, γειτονικές της μεσογειακές χώρες για να δοθεί και έτσι ένα στεναρό μήνυμα ότι είμαστε διατεθειμένοι να φερθούμε στη Λιβύη ως ισότιμο εταίρο με αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό. Ευχαριστώ. Τροπόφιλε. Θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής, είπα της εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, τον κύριο Ντογκέλεβιτς να πάρει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πω ότι η συζήτηση η σημερινή δείχνει ότι η ευρωπαϊκή μας στρατηγική αλλά και η στρατηγική της διεθνούς κοινότητας τους τελευταίους μήνες για τη Λιβύη είχε θετικά αποτελέσματα. Και πραγματικά θεωρώ ότι η Λιβύη είναι ένα σημαντικό εγχείρημα που αποδεικνύει ότι η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική μπορεί να λειτουργήσει. Περάσαμε λοιπόν τις εξετάσεις μας με επιτυχία, θεωρώ, στον τομέα αυτό. Η σημερινή συζήτηση δείχνει ότι η Λιβύη δεν είναι μια απόμακρη χώρα στην οποία πολεμούν οι άνθρωποι. Είναι μια πολύ σημαντική χώρα, σημαντική για την κοινή γνώμη στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια χώρα στην οποία οι Ευρωπαίοι εμπλέκονται και παρακολουθούν τα γεγονότα. Γι' αυτό και έχουμε επιπρόσθετη ευθύνη εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι συμβαίνει στη χώρα αυτή και πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη το καθήκον μας που είναι η στήριξη του λαού της Λιβύης με αυτήν την νέα ελευθερία στην οποία ζουν. Η συζήτηση σήμερα έδειξε επίσης ότι όλες οι προσπάθειές μας για να βοηθήσουμε τη Λιβύη θα πρέπει να στηριχθεί και από τις μη κυβερνητικούς οργανισμούς και όλους αυτούς οι οποίοι μπορούν να παίξουν ένα ρόλο στην ανοικοδόμηση της Λιβύης. Θα στηρίξουμε λοιπόν όλες αυτές τις προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις πτυχές της ανοικοδόμησης. Θα ήθελα επίσης να πω ότι πολλοί ομιλητέ μίλησαν για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον κίνδυνο να συνεχιστούν αυτές οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρετε όμως ότι είπα ότι εκπρόσωπος έχει εκφραστεί σαφέστατα για το θέμα αυτό. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την ευρωπαϊκή αξιολόγηση της κατάστασης και βεβαίως μια πολύ σημαντική ευθύνη και για την μεταβατική κυβέρνηση για τον έλεγχο της κατάστασης διότι εκεί θα πρέπει να παρακολουθήσουμε ότι όλα τα διεθνή πρότυπα τηρούνται και ότι οι κινήσεις που έγιναν μέχρι τώρα είναι οι σωστές. Και αυτό από τις δύο πλευρές. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βρίσκεται στην καρδιά της ευρωπαϊκής πολιτικής έναντι της Νέας Λιβύης. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα εδώ να σταματήσω. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και βεβαίως περιμένουμε με ανυπομονησία το ψήφισμά σας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Η συζήτηση κηρύσσεται πέρα το θύσα. Θέλω να σας ενημερώσω ότι το Προεδρείο έλαβε έξι προτάσεις ψηφίσματος και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι δήλωση